Το θέμα είναι τώρα η δήλωση της ε, Κομισιόν για την υδροηλεκτρική ενέργεια. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ που δίνετε στην Κομισιόν την ευκαιρία να κάνουμε μια ανακοίνωση για το θέμα της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Πρώτα απ' όλα, 40% της ανανεώσιμης παραγωγής ενέργειας είναι υδροηλεκτρική. Οπότε είναι η πρώτη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και θα συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Καθώς πλήρει τους τρεις όρους της ασφάλειας, της εφορίας και της ανταγωνιστικότητας. Η Κομισιόν έχει στόχο να μεταχειριστεί ισότιμα όλους τους παραγωγούς ενέργειας όσον αφορά την πρόσβαση στα, στις υποδομέ. υποδομές. Βεβαίως αυτό σημαίνει πως θα ωφεληθούν και οι τοπικές κοινότητες θα έχουμε εισαγωγή της υδροελεκτρικής ενέργειας στην αγορά και βέβαια θα ωφεληθούν και οι καταναλωτές. Η Κομισιόν γνωρίζει τις οικονομικές, νομικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής. Τα κράτη-μέλη επί της αρχής είναι ελεύθερα να σχεδιάσουν τα μοντέλα τους για την εκμετάλλευση των υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Δεν αμφισβητούμε την αρμοδιότητα των κρατών μελών να επιβάλλουν υποχρεώσεις ε, όταν παραχωρούν τέτοιες εγκαταστάσεις ή συμβόλαια εκμετάλλευσης μπορούν να λάβουν υπόψη όλα τα θεμητά συμφέροντα. Θα πρέπει όμως να σέβονται το σχετικό ευρωπαϊκό δίκαιο. Παραδείγματο το μέλος αποφασίζει να εκμεταλλευτεί τα εργοστάσια αυτά θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες δημοσίων προμηθειών. Το θέμα δεν είναι απλά ζήτημα όρων ανταγωνισμού αλλά και ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στο πλαίσιο αυτό οι κανόνες δημοσίων προμηθειών παραβιάζονται όταν παρατείνεται η αρχική σύμβαση παραχώρησης εκτός εάν αιτιολογηθεί αυτό σωστά. Το ισχύον κοινοτικό δίκαιο μπορεί να διαφέρει αν δεν αποκλείεται η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας ρητά από αυτό. Και θα πρέπει οι παραχωρήσεις και οι σχετικές συμβάσεις να σέβονται το ευρωπαϊκό δίκαιο όπως την οδηγία παραγωγής ηλεκτρισμού. Μάλιστα, οι διαδικασίες διαγωνισμών για συμβάσεις παραχώρησης είναι πάρα πολύ σημαντικές για να λειτουργεί σωστά η αγορά ενέργειας. Τέλος, όταν γίνονται τέτοιες συμβάσεις παραχώρησης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. Όταν λοιπόν δίνονται συμβάσεις παραχώρησης σε μια δημόσια επιχείρηση με κυρίαρχη θέση μπορεί να παραβιάζονται οι κανόνες του ανταγωνισμού, να δημιουργούνται άνισες συνθήκες και να ε, δίνεται η δυνατότητα σε μια δημόσια εταιρεία με κυρίαρχη θέση να την διατηρήσει. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούμε να μιλάμε ακόμα και για κρατικές ενισχύσεις αν μιλάμε για παραχώρηση κρατικών πόρων. Έχουν δοθεί λοιπόν κάποια πλεονεκτήματα σε κάποιες εταιρείε κάτι το οποίο οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Οι συμβάσεις λοιπόν παραχώρησης ε, μπορεί να σημάνει κρατικές ενισχύσεις εάν πρώτον έχουμε κρατικούς πόρους, π.χ. κρατικά έσοδα, τέλη, τα οποία θα, θα μπορούσαν να επιβληθούν. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει ένα επιλεκτικό πλεονέκτημα σε κάποιες εταιρείε έναντι των ανταγωνιστών τους στη συγκεκριμένη αγορά ηλεκτρισμού. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρχει κάποια στρέβλωση του ανταγωνισμού, κάτι το οποίο είναι πιθανόν καθώς ε, πωλείται ο ηλεκτρισμός ε, μεταξύ των κρατών μελών σε ανταγωνιστικές αγορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Συνεχίζεται η συζήτηση για την υδρολητική ενέργεια. Οι πολιτικές ομάδες έχουν τον λόγο. Κύριος Ταγιάννη, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο τομέας της υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι ζωτική σημασία για την ενεργειακή ένωση. Όμως, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι παραχωρήσεις δεν είναι ενιαίο στην Ευρώπη. Σε ορισμένες χώρες μπορούν να ανανεωθούν συμβάσεις παραχώρησης. Αλλού δεν υπάρχει κανένα χρονικό όριο στη διάρκεια μιας σύμβασης παραχώρησης. Πολύ μεγάλες διαφορές δηλαδή και όλα αυτά επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της αγοράς μας. Πρέπει να θεσπίσουμε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ίσους όρους πρόσβασης στους πρωταγωνιστές της αγορές. Αν θέλουμε δηλαδή να έχουμε ισότιμο ανταγωνισμό. Η συζήτηση προέκυψε από το ερώτημα περί του κατά πόσο θα εξασφαλίσει αυτές τις συνθήκες η Κομισιόν στην αγορά. Πώς θα λάβει υπόψη της δηλαδή τις ε, διαφορετικές ε, συμβάσεις παραχώρησης ανά την Ευρώπη. Πρέπει η Κομισιόν να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο, κύριε Επίτροπε, όχι μόνο για τους σκοπούς του ισότιμου ανταγωνισμού, του θεμητού ανταγωνισμού, αλλά και για να ληφθούν υπόψη, όπως είπα, τα καθιστώρα παραχώρησης στον τομέα. Όλα αυτά εν τέλει υπονομεύουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Η κάθε εταιρεία βεβαίως προστατεύεται δικά της συμφέροντα. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε άλλε επιχειρήσει, κυρίω μικρομεσαίε επιχειρήσεις. Θα χαθούν θέσεις εργασία. Θα έχουμε απώλειες στον τομέα τη ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λέω ότι μία επιχείρηση φυσικά είναι υπεύθυνη για όλα αυτά, για το μέλλον του τομέα. Ε, πάντως, κύριε Επιτροπέ, μέσω ημών θέλω να καλέσω την Κομισιόν να αναλάβει πρωτοβουλία πρέπει να υποστηρίξουμε τον τομέα. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο Από τους σοσιαλιστές, η κυρία Τόγια, Ιτρελετά. Κύριε Πρόεδρε, ο τομέα είναι σημαντικότατο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Συμβάλλει στην οικονομία, το συνολικό του τομέα, ο κύκλος εργασιών είναι ίδιο με το ΕΠ της Σλοβακίας. Λοιπόν, Ξεχάσαμε τα εμπόδια και τα προβλήματα του τομέα δυστυχώς. Ξεχάσαμε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές από χώρα σε χώρα όσον αφορά τις παραχωρήσεις. Μιλούμε και για την αγορά ηλεκτρικού ρεύματο. Οι διαφορές λοιπόν αυτές σημαίνουν και στρέβλωση του ανταγωνισμού και λιγότερη ανταγωνιστικότητα, λιγότερες επενδύσεις και όχι βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων. Η Κομισιόν έχει περιπέσει αντιφάσεις, νομίζω, στην υλοποίηση της πολιτικής της. Η Γενική Διευθύνση Ανταγωνισμού κάνει το α, αλλά κάνει και το αντίθετό του, υιοθετώντας κάθε φορά διαφορετικές οπτικές γωνίες. Όλα αυτά είναι λίγο ατάκτως ερημένα. Σημαίνουν λοιπόν παράδοξα, κάποιες χώρες την χάνουν δυσμενέστερη μεταχείριση και όλα αυτά διότι δεν σπεύσαμε να απελευθερώσουμε πώς έπρεπε την αγορά αυτή. Υπάρχουν λοιπόν συμβάσει παραχώρηση χωρί χρονικό όριο. Αυτό παραλαμβάνω σημαίνει μικρότερη ανταγωνιστικότητα. Και σε κάποιε άλλε χώρε, κάποιε άλλε χώρε, τι τρέχουμε στα δικαστήρια. Σα ζητώ λοιπόν, κύριε Επίτροπε, να επέμβετε. Όχι, όχι εσεί προσωπικά, αλλά κάποιο συνάδελφο στο Κολέγιο των Επιτρόπων να θεσπίσει ενιαίου κανόνε για όλου. Αλλιώ έχουμε στρέβλωση του αιωνισμού. Χρειαζόμαστε μια διαφορετική προσέγγιση επίση στι περιπτώσει παραβίαση. Χάνουμε την αξιοπιστία μα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα για διαφορετικέ χώρε, σε διαφορετικέ περιπτώσει. Δεν είναι αυτή η λύση για την Ενεργειακή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κ. Σελίμοβιτ, εκ μέρου των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ από όταν η Κομισιόν συνέταξε μια στρατηγική σχετικά με το θέμα αυτό για το 2015. Το σκεπτικό ήταν ότι όλοι θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή παροχή ενέργειας. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να έχουμε και την υδροηλεκτρική ενέργεια εδώ, γιατί 60% των ΑΠΕ είναι υδροηλεκτρική ενέργεια, ενώ το 2006 πριν 10 χρόνια ήταν μόλις 6%. Οπότε μπορούμε πέρα από την καλύτερη διαχείριση των πόρων να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε την υδροηλεκτρική ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται ακόμα. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες π.χ. στην Αλβανία, Βοσνία κτλ. που απέχουν ακόμα πολύ από το να επιτύχουν τα ποσοστά που θα μπορούσαν. είναι λοιπόν απλά θέμα διασύνδεσης και καλύτερων ρυθμίσεων. Πρέπει να δούμε και την γειτονιά μας για να επιδευτεί ο στόχος της Ενεργειακής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να ακολουθούμε και τους ε, κανόνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υδροελεκτρική ενέργεια. Σας ευχαριστώ για την QNGL. Η κυρία Λόπες Μπερμεχό, για ένα μισή λεπτό. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε επειδή τις δύο φορές που γραπτός ρώτησα για τις παραχωρήσεις προς τις επιχειρήσεις ενέργεια ενέργειας Πανικές, Η Κομισιόν μου δεν είχε πληροφορίε. Τι γίνεται με τα θέματα ανταγωνισμού. Οι πληρωμές προ αυτές τι επιχειρήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ το κόστο των επενδύσεων και έχουν καταγραφεί παρατυπίε όπως καθυστερήσεις ή επιστροφές των κονδυλίων στο δημόσιο τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένη απάντηση για αυτή την κατάσταση. Γιατί μου φαίνεται παράδοξο που η Κομισιόν που είναι τόσο ενεργή σε άλλου ε, τομεί φαίνεται να παραγνωρίζει και να αγνοεί τη βλάβη προ του καταναλωτέ από τι επιχειρήσει του τομέα. Και όχι μόνο ε, στο θέμα τη ρύθμιση των τιμών. Οι κυρώσει και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στην Ισπανία για τις τιμές στην ουσία βοηθούν τους μεγάλους παραγωγούς. Αυτό καταγγείλουμε εδώ και πολύ καιρό. Σας το ρωτώ αυτό με την πεποίθηση ότι η ενέργεια αυτή διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στο θέμα και στον κλάδο της ενέργειας σε σχέση και με άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν αυτό που κάνουμε να λαμβάνει υπόψη του το γενικό συμφέρον και θα πρέπει να δίνουμε και σημασία στην διατήρηση των οικοσυστημάτων και στην προστασία του γεωργικού τομέα. Οπότε εδώ χρειάζεται καλύτερο συντανισμό μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και των υπευθύνων. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι ακριβώς θέλει να κάνει η Κομισιόν και για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μισελ Ριβαζή, εξ ονόματο των Πρασίνων. Έχετε το λόγο για να το παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η ηλεκτρική ενέργεια νομίζω ότι αποτελεί πραγματικά μια κληρονομιά για κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Μας επιτρέπει να συμπληρώσουμε την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά συμβάλλει και σε θέματα που αφορούν το τοπίο. Δεν έχουμε να κάνουμε λοιπόν μόνο με την με την ενέργεια αλλά και με στρατηγικά ζητήματα που αφορούν τον πληθυσμό, ιδιαίτερα αυτό που μένει κοντά σε παράκτητες περιοχές. Στα πλαίσια λοιπόν των παρηχωρήσεων, το, θέμα, το θέμα δεν είναι κατά πόσο ο φορέας θα είναι ιδιώτης ή το κράτος. Το ζήτημα είναι ακριβώς ποια προσθέμενη αξία ένας νέος εντολογοδόχος θα ποια αξία θα έχει αυτός και πώς θα δουλέψει. Τώρα για τις ε, παραχωρήσεις θα πρέπει να, δούμε ακριβώς πώς γίνονται. Ο κατακαιρματισμός τους και η έλλειψη σφαιρικής προσέγγισης θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Τα ατυχήματα θα έπρεπε να αποφευθούν χάρη στο συντονισμό που θα πρέπει να υπάρχει. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι απλή. Η Κομισιόν θα προωθήσει τις συμβάσει παραχώρησης αναγκατάσταση ή θα λάβει υπόψη της γενικότερα τα στοιχεία του οποίου ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εκ μέρου του ευθυντητή ο κύριος Χέλμαρ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συχνά είπα ότι είμαι κατά της ηλιακής και αιωλικής ενέργειας εδώ. Με χαρά λοιπόν βρίσκω μια ΑΠΕ την οποία στηρίζω, η οποία είναι προβλέψιμη, είναι αξιόπιστη, είναι φτηνή. Χρειάζεται λίγη συντήρηση και λειτουργεί χωρίς επιδοτήσεις και μάλιστα σε πολλές, από πολλές απόψεις είναι το τελείως αντίθετο της αιωλικής και της ηλιακής πάνω στις οποίες έχουμε ξοδέψει τόσα χρήματα τα τελευταία χρόνια αυξάνοντας τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και ε, οδηγώντας χώρες να αφήνουν την Ενώση. Βέβαια το πρόβλημα είναι η διάθεση της θελακτικής ενέργειας η οποία περιορίζεται ανάλογα με την τοποθεσία και την τοπογραφία. Τώρα εμείς ακούμε κλήσεις για εναρμόνιση των κανόνων όσον αφορά τις, ε, την παραχώρηση των αδειών. Εμείς είμαστε κατά οποιασδήποτε κίνηση για εναρμόνιση. Οι πόροι, οι υδροελεκτρικοί στην χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελούν εθνικό πόρο και θα λάβουμε μέτρα σημαντικά για να προστατεύσουμε αυτούς τους πόρους από τις Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Καρίνς, ένα μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, το καμπανάκι χτυπάει, μπαίνουν οι δύο μποξέρ ε, στο ring, ο ένας έχει το ένα δε, χέρι δεμένο πίσω από την ε, πλάτη του. Αν βλέπαμε κάτι τέτοιο θα λέγαμε ε, είναι αδικία, δεν είναι σωστός αγώνας αυτός, ούτε δίκαιος ανταγωνισμός. Τι βλέπουμε όμως τώρα στην αγορά της ενέργειας και ειδικά της υδροηλεκτρικής, βλέπουμε σε διάφορες χώρες διαφορετικούς κανόνες για την υδροηλεκτρική ενέργεια το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι το παραγόμενο ρεύμα περνάει ελεύθερα τα σύνορα και πωλείται σε μια κοινή αγορά. Έτσι όμως τρευλώνεται ο ανταγωνισμός γιατί η παραγωγή γίνεται με διαφορετικές συνθήκες στην ε, κάθε χώρα. Οι επαιτήσει ε, για τις επενδύσεις. Ε, όλα αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Όμως το ρεύμα είναι σε μία ενιαία αγορά. Σαν έναν μποξέρ δηλαδή, ο οποίος είναι αναγκασμένος να παίζει με το ένα χέρι δεμένο στην ε, πλάτη του απέναντι σε ένα που έχει τα χέρια του ελεύθερα. Αν είναι να έχουμε δίκαιο ανταγωνισμό και σωστή αγορά ενέργεια στην Ευρώπη, πρέπει και οι δύο μποξέρ να έχουν τα χέρια τους ελεύθερα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ζαν Πολ Τζένανο για ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, με την προφορική ερώτηση θέλησα να επιστήσω την προσοχή της Κομισιόν στον σημαντικό ρόλο της μορφής αυτής της ενέργειας. Διότι αποτελεί ανανεώσιμη και αποθηκεύσιμη μορφή ενέργειας, συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών, διοξιδίου του άνθρακα, συμβάλλει στην ασφάλεια, στην ενεργειακή ασφάλεια και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά δεύτερο λόγο, ο τομέα της υδροελεκτρικής ενέργειας συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τοπίου και στη διατήρηση θέσεων εργασίας στο τοπικό επίπεδο. Σχετίζεται όμως με τη γεωργία, με το πόσιμο νερό, με την αυσιπλοεία, με τον τουρισμό, με την ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω την προσοχή της Κομισιόν στην ανάγκη να διελευκανθεί και να διευκρινιστεί η κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη των κανονισμών που διέπουν τον τομέα. Όπως έδειξε και πρόσφατη μελέτη, το να ανοίξουμε τον τομέα στον ανταγωνισμό θα έχει επιπτώσει σε ορισμένε χώρε μέλη, όχι όμω σε άλλε. Κινδυνεύουν όμω τα οικοσυστήματα. Γι' αυτό α προσέξει η Κομισιόν να καταλήξει γρήγορα σε κάποια συμπεράσματα, προσέχοντα όμω να μην ανοίξει την πόρτα σε μια πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών που εν τέλει θα πλήξει την αγορά ενέργεια στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σέσκουν Βιλμπάου βαραντικά. Πρώτα ευχαριστώ. Ναι, Επίτροπε, η Ευρώπη είναι μια από τις περιοχές ε, παγκοσμίω με μεγαλύτερη παρουσία υδροελεκτρικής ενέργειας, παρόλο που πολλές από τις εγκαταστάσεις ε, παρουσιάζουν ευκαιρίες τεχνολογικής βελτίωσης αφορά την κατεστημένη ισχύ. Και ε, τη μορφή ΑΠΕ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη λόγω της δυνατότητας αποθήκευσης, κάτι το οποίο επιφέρει σταθερότητα στην αγορά, τη στιγμή που κάποιες άλλες πηγές ΑΠΕ παρουσιάζουν αυξημίωση. Γι' αυτό ακριβώς η έμφαση στην τρολεκτρική ενέργεια πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ένεση. Αυτό όμως ως δέσμευση αντιβαίνει σε αυτό τον λαβύρινθο νομοθεσίας της ε, Ένωσης Έχουμε πολλά καθεστώτα, κανόνες κλπ. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να υπάρχουν διοικητικοί και νομικοί κανόνες που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια δικαίου και την ασφάλεια των επενδύσεων. Σε κάποιες χώρες όπως η Ισπανία οι επιχειρηματίες έχουν εγκλωβιστεί σε μια διαδικασία επιδότησης των ΑΠΕ που είναι ένα παράδειγμα του κακών επιπτώσεων που έχουν οι ευρωπαϊκές στρατηγικές στους παραγωγούς και στους καταναλωτές ιδιαίτερα όσον αφορά την προσφορά ενέργειας. Γι' αυτό ακριβώς κύριε Επίτροπε θα ήθελα να μάθω πότε ακριβώς θα σταματήσει να υπάρχει ανασφάλεια και πότε ακριβώς θα μπορέσουμε με τους παραγωγούς στο πλαίσιο των σωστών παραχωρήσεων να θεσπίσουμε επιτέλους τα σωστά κίνητα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Γκροστέτ. Γκροστέτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. 16% της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στον κόσμο προέρχεται από την υδροελεκτρική ενέργεια. Είναι η τρίτη πηγή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Πάρα πολύ σημαντικό. Ζωτική σημασία λοιπόν για την Ευρώπη. Υποστηρίζει χιλιάδες θέσεις εργασίας επιτόπου. Υποστηρίζει το περιβάλλον και στα βουνά και στις παιδιάδες. Οι παλιοί μήλοι, τα φράγματα, αποτελούν μέρος της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Πρόκειται για ενέργεια η οποία δεν παράγει διοξίδιο του άνθρακα βεβαίω, κάτι το οποίο συνάδει με τους ενεργειακού και περιβαλλοντικού μας στόχου. Όμως, δεν πρόκειται μόνο για τι ανανεώσιμε πηγέ. Είναι ενέργεια η οποία είναι και αποθηκεύσιμη. Η απελευθέρωση τώρα δεν πρέπει να γίνει με τρόπο βίαιο και βιαστικό. Πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και η Γαλλία ε, έκαναν πολλές προσπάθειες και δυστυχώς τώρα τις αγνοούμε. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην σταματήσουμε τις επενδύσεις στον τομέα. Το μήνυμα που στέλνει σήμερα στους επενδυτές η Κομισιόν δεν ήταν φοβούμε αρκετά θετικό. Η αλήθεια είναι ότι σε μερικά μελη ο ανταγωνισμός ε, δεν υπάρχει, είναι πολύ περιορισμένος κάποιοι που θέλησαν να επενδύσουν αποθαρρύνθηκαν. Λοιπόν, πώς σκοπεύει η Κομισιόν να ευνοήσει την ανάπτυξη του τομέα. Η να το ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη, κυρίως στις ορεινές ζώνες. Ευχαριστώ πολύ. Σον Κελή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που γίνεται αυτή η συζήτηση έστω και τόσο αργά για το θέμα των ΑΠΕ. Στην υδροηλεκτρική ενέργεια έχουμε έναν κλάδο 100 ετών με πάρα πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα από οποιαδήποτε άλλη πηγή παραγωγής ενέργειας. Μιλάμε για μεταξύ 80 και 90%. Μια καθαρή πηγή ενέργειας που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους κλιματικούς στόχους. Με 390 τεραβάτα εγκατεστημένη ισχύ είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο σημαίνει 24 δισεκατομμύρια ευρώ εξοικονόμηση από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Η Ευρώπη λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάει προς τη ΣΑΠΕ όχι μόνο για την κλιματική αλλαγή αλλά και για να μειώσουμε 400 δις που δίνουμε για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων κάθε χρόνο. Η υδροελεκτρική ενέργεια λοιπόν είναι ιδανική καθώς όταν λάμπει ο ήλιος ή φυσάει ο αέρας μπορούμε να γεμίσουμε τους ταμιευτήρες για τις στιγμές που δεν θα φυσάει ο αέρας ή θα λάμπει ο ήλιος. Και βεβαίως μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική αποθήκευση ενέργειας και η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η μοναδική τέτοια τεχνολογία μεγάλης κλίμακας που είναι ήδη σήμερα διαθέσιμη. Μας επιτρέπει λοιπόν να έχουμε αποθήκευση της ενέργειας και ελαστικότητα στο σύστημα. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα νέο σχεδιασμό της αγοράς για να υπάρξει ακριβώς εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων της. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μασιμιλιάνο Σαλίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σκέψεις συγκεκριμένες, για έχει περάσει η ώρα. Να είμαστε ακριβείς και απλοί. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πολλοί τρόποι παραχώρησης στα υδροελεκτρικά. Υπάρχουν χώρες που δεν κάνουν διαγωνισμούς, άλλες που κάνουν διαγωνισμούς, αλλά μετά τους διαγωνισμούς αυτούς έχουμε μια παράταση της παραχώρησης χωρί να υπάρξει νέο διαγωνισμό. Και υπάρχουν χώρε που γίνονται τακτικά διαγωνισμοί, όπου μετά την περίοδο παραχώρηση έχουμε και πάλι διαγωνισμό. Σε αυτέ τι χώρε λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα οικονομικό και νομικό. Και από ό,τι φαίνεται η Κομισιόν δεν το έχει λάβει υπόψη τη σοβαρά. Επειδή ακριβώ αν η απόσβεση των επενδύσεων διαρκέσει για περισσότερο χρόνο από την παραχώρηση, τότε είναι φυσιολογικό μετά την παραχώρηση να υπάρξει μια υπολείπουσα απόσβεση. Οπότε αυτός που θα κερδίσει το διαγωνισμό θα πρέπει να πληρώσει ακριβώς την υπολείπουσα απόσβεση στον προηγούμενο παραχωρησιούχο. Πολύ απλό αυτό. Η Κομισιόν όμως δεν το έχει καταλάβει. Και έχει παρενέβει τιμωρώντας τις χώρες που εφαρμόζουν αυτόν τον κανόνα, που είναι ένας κανόνας διαφάνειας και ανταγωνισμού. Οπότε θεωρώ ότι είναι σωστό να υποστηρίζουμε αυτούς που κάνουν τις επενδύσεις, αλλά είναι σωστό εξίσου να υποστηρίζουμε αυτούς που μέσω ελεύθερου ανταγωνισμού αποφασίζουν να διασφαλίσουν στους ε, πιθανούς επενδυτές τους ε, κανόνες της αγοράς. Είναι καλό λοιπόν να το αντιληφθεί αυτό η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Σαλίνη. Ο κύριος Τζοβάνι Λαβία. Παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος στα Ιταλικά. Κύριε Επίτροπε, σήμερα συζητάμε ένα θέμα τεράστιας ε, σημασίας. Στο Παρίσι συμφωνήσαμε μία παγκόσμια δέσμευση για μία σημαντική μείωση ώστε να αντιμετωπιστεί κλιματική αλλαγή. Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε νέες μορφές ενέργειας, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ενέργεια με χαμηλό αντίκτυπο άνθρακα. Τα υδροελεκτρικά αυτό ακριβώς είναι και μας επιτρέπουν να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία στην διαδικασία παραγωγής. Η υδροελεκτρική όμως ενέργεια στην Ευρώπη απειλείται επειδή φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρχουν επαρκείς επενδύσεις και συντήρηση των ε, προχωρών εγκαταστάσεων, αλλά ακριβώ έλλειψη πλαισίου. Κάποιο μίλησε για ανταγωνισμό. Το ζήτημα είναι πιο σοβαρό. Δεν γίνεται στην ίδια, την, στην ίδια αγορά, στην ενιαία αγορά ενέργειας που επιθυμούμε στην Ευρώπη, να υπάρχει καποιο ο οποιο διατηρεί προνομιακές θέσεις, απολαμβανοντα ιδιαίτερων προνομίων που έχει στι εθνικέ αγορές και μετά έχει και την ευκαιρία να πάει σε άλλες αγορές. Ενώ για άλλους οι εθνικές αγορές είναι ανοιχτές και δεν έχουν δυνατότητα να πάνε παραπέρα. Γι' αυτό ακριβώς Επίτροπε χρειαζόμαστε ένα νομοθετικό πλαίσιο νέο και ομοιογενές το οποίο θα είναι ισότιμο για όλους, θα διασφαλίσει τον οργανισμό και θα ε, προωθεί τις επενδύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λαβία, λέγει ο στα τελικά. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε χρόνο για διαδικασία κατσδιάη. Μισελ Ντάντεν, παρακαλώ. Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, το φράγμα παράγει ρεύμα. Όμως, είναι και θέμα διαμόρφωσης του τοπίου. Κάνει το τοπίο πιο ελκυστικό ένα εργαλείο αν θέλετε και είναι και ένα θέμα το οποίο αφορά τον τοπικό πληθυσμό. Οι διαφορές μεταξύ των απόψεων εντός της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας ε, δεν μπορούν να συνεχιστούν. Ας ε, συμφωνήσουμε επιτέλους και ας βάλουμε μια τάξη στην ενεργειακή μας πολιτική και στην πολιτική ανταγωνισμού. Το θέμα της εκμετάλλευσης και της αξιοποίησης των ε, εγκαταστάσεων αυτών πρέπει και αυτό να ρυθμιστεί. Πρέπει κάτι να κάνουμε μια νομοθεσία που να μπορεί να εφαρμοστεί παντού σε όλες τις χώρες προς μια Ευρώπη της ενέργειας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο υδροηλεκτρικός τομέας παράγει 15 με 20% του ρεύματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όπου απασχολεί περί τους 80.000 εργαζόμενους. Είναι και θα παραμείνει για αρκετά χρόνια η πρώτη από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συνεπώς διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων του Horizon 2030 δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι στο ξεπούλημα της ΔΕΗ στην ελλάδα που επιχειρεί η τρόικα και οι μνημονιακές κυβερνήσεις τα υδροηλεκτρικά φράγματα αποτελούν πρώτης τάξεως φιλέτα για τους υποψήφιους επενδυτές. ο υδροηλεκτρικός τομέας ωστόσο έχει ανάγκη τις απαραίτητες επενδύσεις για να διατηρηθεί ανταγωνιστικός επενδύσει στην καινοτομία και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του υπάρχοντος δυναμικού αλλά και στη διαχείριση και πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υδροηλεκτρικών φραγμάτων αυτές οι επενδύσεις δεν θα γίνουν ποτέ από τους ιδιώτες που προσβλέπουν στο άμεσο και βραχυπρόθεσμο κέρδος. τα ελληνικά υδροηλεκτρικά φράγματα πρέπει λοιπόν να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο μακριά από το χέρι της τρόικας και των δανειστών με μόνο γνώμονα το όφελος του ελληνικού λαού και την ευημερία του. ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, ο κύριος Άντριο Κάιτης, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ για την πολύ χρήσιμη αυτή συζήτηση. Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι σημαντική απέ και ένα σημαντικός κλάδος της οικονομίας της Ένωσης. Η ποικιλομορφία όμως ε, των ρυθμιστικών καθεστώτων είναι ένα γεγονός είναι σημαντικό οι συμβάσεις παραχώρησης να σέβονται το υφιστάμενο ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να επιβλέπει την εφαρμογή των κανόνων. Αυτό είναι σύμφωνα με τους κανόνες της Ενεργειακής Ένωσης για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά. Και βεβαίως να υπάρχει ε, ενεργειακή ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εξετάζουμε τι συμβάσεις παραχώρησης σε κάποια κράτη-μέλη. Έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάση και μπορεί να ξεκινήσουμε και άλλες εάν δούμε πώς έχει υπάρξει παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου και της οδηγίας περί παραχωρήσεων, περί υπηρεσιών και ανταγωνισμού. Και κάποιοι ανέφεραν το ότι η Κομισιόν δεν συνεργάζεται. Όχι. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Ενέργειας ε, και Ανταγωνισμού. Υπάρχει ίση μεταχείριση των κρατών μελών επίσης. Και η Κομισιόν αυτή τη στιγμή εξετάζει διάφορα εθνικά αριθμιστικά καθεστώτα και όπου είναι αναγκαίο θα δράσει για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Σας ευχαριστώ. Mm, Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρέμβαση.